με ανάπτυξη και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και ότι αυτά είναι εξίσου σημαντικά επιδιώκοντα τα συμφέροντα τα εμπορικά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπέρμπερ. Για ένα λεπτό ο κύριος Ενά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι.